άρθρου 166 του κανονισμού αποφάσισα να επιβάλλω ποινές στον ε, ε, κύριο Κόρβιν Μίκη και κύριο Μπουνάνο για την τεραχή τη σωστή ε, διενέργηση τη συνεδρίαση τη 7η Ιουλίου και 8η Σεπτεμβρίου, καθώ και τη 6η και 7η Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν για 10 ημέρες δεν θα έχουν τις δραστηριότητέ του καθώ και την αποζημίωσή του στην ημερήσια. Και για 10 λοιπόν ημέρε θα αποσχούν από τι δραστηριότητε ε, του Κοινοβουλίου και όλων των σχετικών οργάνων και την απόφαση αυτή την κοινοποίησα στα μέλη αυτά την προηγούμενη εβδομάδα και την πρώτη τελευταία εβδομάδα ο κύριος Κόρβιν Μίκεν και ο κύριος Μπουνάνο σύμφωνα με τον άρθρο 167 υπέβαλαν ιστορική προσφυγή κατά, την απόφαση, κατά τις απόφασεις αυτής και το Προεδρείο θα εξετάσει σήμερα το βράδυ τις δύο αυτές προσφυγές και θα λάβει τη σχετική απόφαση από πλευρά της διαδικασία. Αυτό σημαίνει το Προεδρείο. Έχετε την δυνατότητα να άρει ή επιβεβαιώσει τις κυρώσεις που επέβαλα την απόφαση του Προεδρείου θα την διαβιβάσουμε άμεσα στους βουλευτές και σε περίπτωση επικύρωσης των αποφάσεών μου θα έχουν άμεση ισχύ οι κυρώσεις. Για αυτό το θέμα επιθυμείτε το λόγο ή για άλλο θέμα, για άλλο ζήτημα. Ε, λίγο αργότερα, λίγο αργότερα αν θέλετε.